στην ψηφοφορία του συνόλου της πρότασης για το διορισμό του κυρίου Αλτζίρτας σε μέτα ως μέλους της Επιτροπής. Υπενθυμίζω ότι αυτός ο Επίτροπος θα αντικαταστήσει την κυρία Γκρίμπο Στάιτε, η οποία εξελέγει πρόεδρος της Λιθουανίας και προς την οποία θα ήθελα να εκφράσω και κάθε ευτυχία, όλες τις ευχές μου και εκ μέρου σας. Ψηφίζουμε μυστικά. Θέτω σε ψηφοφορία λοιπόν την πρόταση απόφασης. Ξεκινάει η ψηφοφορία.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 Ψήφι υπέρ 347 ψήφι, κατά 47, αποχές 67. Επομένως, η πρόταση εγκρίνεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε... Α, καταρχάς ξέχασα να πω καλή επιτυχία στον καινούργιο επίτροπο. Θα ψηφίσουμε τώρα την πρόταση απόφασης για την έγκριση του διορισμού του Πάουελ Σαμέκη μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο, στη θέση της κυρίας Ντανούτα Χούμπνερ που είναι συνάδελφός μας τώρα. Θα θυμάστε ότι ήταν υπεύθυνη για την περιφερειακή πολιτική και την πολιτική συνοχής. Θα ψηφίσουμε μυστική ψηφοφορία και εδώ. Θα ήθελα να ψηφίσουμε λοιπόν την πρόταση απόφασης έναρξη ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορία. Ψήφισαν 474 βουλευτές, 360 υπέρ, 80 κατά, 34 αποχές. Εγκρίνεται η πρόταση. Καλή επιτυχία. Και τώρα θα ψηφίσουμε την πρόταση για την έγκριση του διορισμού του Κάρελ Ντεγκούκτα μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη θέση του Λί Μισελ, που και εκείνο έγινε τώρα Ευρωβουλευτής και συνάδελφός μας. Θα ήθελα να ψηφίσουμε αυτή την πρόταση, επίσης με μυστική ψηφοφορία. Έναρξη ψηφοφορίας παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Ψήφισαν 472, 385 υπέρ, 53 κατά, 34 αποχές. Εγκρίνεται και αυτή η πρόταση. Καλή επιτυχία στον νέο επίτροπο λοιπόν. Bene. Adesso Τώρα Για μισή ώρα έχουμε τις παρεμβάσεις ε, του ενός λεπτού. Υπάρχει ένας τεράστιος κατάλογος από αιτήματα. Υπάρχει τεράστια βούληση για συμμετοχή που δείχνει και τη σημασία και το ενδιαφέρον στη δουλειά του Κοινοβουλίου. Φυσικά δεν μπορώ να δώσω το λόγο σε όλους όσοι τον ζήτησαν. Γιατί σε αυτήν την περίπτωση θα έπρεπε να έχουμε στη διάθεσή μα μία μισή ώρα. Ενώ έχουμε στη διάθεσή μα μόνο 30 λεπτά. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Κέλλη. Σον Κέλλη.